Ε, πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ κυρία Παναγιώτοβα και του Συμβούλιο που εκπροσωπείτε. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 2 του κανονισμού έχω λάβει ένα αίτημα από την Επιτροπή Γυναικών ε, για να γίνει διερευνητική γνωμοδότηση από την ΕΟΚΕ για ε, διακρίσεις ε, με βάση το φύλλο στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. Αν δεν διαφωνεί μια πολιτική ομάδα ή ε, κάποια μέλη, αριθμός μελών που απαιτούνται εντός 24 ωρών, θα εγκριθεί αυτό το αίτημα, αλλιώς θα τεθεί σε ψηφοφορία. Και τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι ανακοίνωση ε, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σχετικά με την ε, απόφαση του δικαστηρίου στην Ισπανία σε σχέση με την υπόθεση Λαμανάδα ή Αγέλη. Thank you, President, honorable member. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Βουλευτέ, κύριε Επίτροπε. Το ότι